Σας ευχαριστώ. Τελείωσε εδώ πέρα η συζήτηση. Η ψηφοφορία αύριο 6 ε, ώρα το απόγευμα. Επόμενο σημείο, έκθεση Μορέιρα για τις οικονομικές και εμπορικές σχέσεις με τις ΗΠΑ. Ο εισηγητής έχει το λόγο για τέσσερα λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι. φτάσαμε σε αυτή την ώρα την νυχτερινή και μιλάω για να καταγραφούν αυτά που λέω. Αυτά έχω να πω παρουσιάζω στην έκθεσή μου για τις εμπορικές και οικονομικές σχέσεις με τις ΗΠΑ, η οποία εγκρίθηκε από την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου με μεγάλη πλειοψηφία. Όσον αφορά τι εμπορικέ σχέσει με τι Ηνωμένε Πολιτείε, πρέπει να πω ότι είμαι εξαιρετικά ικανοποιημένο από την ουσία τη έκθεση. Γιατί καταρχήν στέλνει μια έντονη, ένα έντονο μήνυμα ε, στήριξη στη βελτίωση των εμπορικών και οικονομικών σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένων Πολιτειών και δεύτερον η έκθεση αναφέρει τις πιο, τα πιο σημαντικά επιθετικά και αμυντικά στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν θέτει προϋποθέσεις για το άνοιγμα των περαιτέρω διαπραγματεύσεων. Η φύση της έκθεσης κυρίως είναι πολιτική. Αυτό το οποίο προσπαθούμε να κάνουμε είναι να στείλουμε ένα μήνυμα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να στηρίξουμε το άνοιγμα των διαπραγματεύσεων για μια εμπορική συμφωνία και για εμπορικά μέσα μεταξύ ευρωπαϊκή Ένωση και Ηνωμένων Πολιτειών με σκοπό τη δημιουργία μιας πραγματικής διατλαντικής αγοράς. Η έκθεση αυτή προσπαθεί να απαντήσει σε δύο βασικά ερωτήματα. Πρώτον, αν υπάρχει συμφωνία εμπορίου και επενδύσεων έχει νόημα αυτό. Ναι, όλοι θα συμφωνήσουν ότι έχει νόημα. Όλες οι έρευνες δείχνουν ότι υπάρχει τεράστια δυνατότητα ανάπτυξης με μια αμοιβαία απελευθέρωση εμπορίου και επενδύσεων από τις δύο πλευρές. Ταυτόχρονα και οι δύο οικονομίες αντιμετωπίζουν παρόμοιες δυσκολίες που μπορούν να αντιμετωπιστούν μάλλον από κοινού παρά ε, χωριστά από τον καθένα. Και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε περαιτέρω ανάπτυξη, κυρίως δεδομένου ότι από κοινού αντι, ε, μπορούμε να ανοίξουμε αγορές όπως η Βραζιλία, η Αργεντινή και η Νότιος Αφρική. Ε, επιπλέον, ο γύρος της Ντόχα για τις πολυμερείς ε, εμπορικές ε, συμφωνίες μάλλον απέτυχε και τώρα μπορούμε να προχωρήσουμε μόνο σε διμερές επίπεδο. Επιπλέον, θα είναι δυνατόν να επιτευχθεί συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών σε λογικό χρονικό διάστημα. Εδώ αναφέρεται ότι αυτό δεν θα είναι εύκολο. Υπάρχουν ε, διαφορετικά συμφέροντα σε σημαντικού τομεί όπως η γεωργία και οι θαλάσσιες μεταφορές. Αυτά είναι δύο από τα παραδείγματα. Υπάρχουν ε, ε, νομοθετικές διαστάσεις όσον αφορά τα πρότυπα για τα αυτοκίνητα. Υπάρχουν και πολιτιστικές διαφορές μεταξύ ΗΠΑ και Ευρώπης. Οι Ευρωπαίοι ενδιαφέρονται πολύ για την αρχή της πρόληψης όσον αφορά τη γεωργία και τη βιομηχανία ενώ οι Αμερικανοί, στους Αμερικανούς αρέσει να λαμβάνουν κινδύνους. Υπάρχουν και προβλήματα με τους γενετικά μεταλλαγμένους οργανισμούς από κάθε πλευρά. Υπάρχουν διαφορετικές απόψεις στο θέμα της χρήσης των ε, κλώνων των ζώων. Ε, είναι δυσκολίες που όμως κατά τη γνώμη μου μπορούν να ξεπεραστούν. Αυτά είναι ε, εμπόδια για την επίτευξη ε, επιτυχημένης ε, εμπορικής συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί πρέπει οι συμφωνίες να καλύψουν όλους τους τομείς και να αφαιρεθούν τα εμπόδια στο εμπόριο σε όλους αυτούς τους τομείς. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να ξεκινήσουμε διαπραγματεύσεις για να μπορέσει να επιτευχθεί μια αποδεκτή συνένεση και στις δύο πλευρές για να μπορέσουμε να επιταχύνουμε το εμπόριο ε, καταργώντας τα εμπόδια όπως είναι τα τεχνικά στάνταρτ. Είναι σημαντικό λοιπόν το κοινοβούλιο αυτό να αντιμετωπίσει με σοβαρότητα την έκθεση και να δώσει ε, ε, ενθάρρυνση και στην Κομισιόν και στο Συμβούλιο για να συνεχίσουν τις συζητήσεις στον τομέα αυτό με τις ΗΠΑ. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ξεκινάει η διαδικασία και έτσι διάει ο κ. Νικολάσιτς. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αυτή είναι μια πολύ θετική είδηση για τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συναλλάσσονται με τις Ηνωμένες Πολιτείες γιατί η θέση τους θα βελτιωθεί. Επειδή θα μπορέσουν να διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας, να, αυξηθούν, να αυξήσουν τις θέσεις εργασίας, να αυξηθεί το εμπόριο και στις δύο πλευρές. Όμως υπάρχουν μια σειρά από θέματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν όπως είπε και ο εισηγητής. Υπάρχουν διαφορές μετα... που αφορούν ε, τεχνολογικά ζητήματα για την αγορά και πώληση αυτοκινήτων για τη χρήση γενετικά μεταλλαγμένων οργανισμών, που είναι ένα ευαίσθητο ζήτημα για τους πολίτες της Ευρώπης. Βεβαίως, οι διαπραγματεύσεις μπορεί να ευοδοθούν. Επίσης, το κρέας από ε, ζώα κλόνους είναι επίσης ένα ευαίσθητο θέμα για μας. Όμως, εν κατακλείδη μπορούμε να πούμε ότι βεβαίως η βελτίωση των εμπορικών σχέσεων μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΗΠΑ για μας είναι απαραίτητη. ευχαριστώ για να ολοκληρωθεί η διαδικασία η κυρία Τσικάου. Οι εμπορικές και οικονομικές σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών στον τομέα των μεταφορών είναι απαραίτητη και χρειάζεται μεταρρύθμιση των διατάξεων για τη συμμετοχή ξένων κεφαλαίων στις αμερικανικές εταιρείες. Ο προστατευτισμός ε, ε, των αμερικανικών αεροπορικών εταιριών και η αδυναμία πρόσβασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ευρωπαϊκών, των ευρωπαϊκών εταιριών στην αμερικανική αγορά, η δυνατότητα καμποτάζ, ε, στις Ηνωμένε Πολιτείε όταν οι αμερικανικές αεροπορικές εταιρείε έχουν τη δυνατότητα καμποτάζ στην Ευρώπη. Πρέπει όλα αυτά να σταματήσουν. Πρέπει να, να αξιοποιήσουμε το σύστημα GPS Γαλιλαίος που θα μας βοηθήσει να αναπτυχθούμε στον τομέα των μεταφορών για να αντιμετωπίσουμε τον ανταγωνισμό. Τώρα χρειάζεται συνεργασία όσον αφορά στις μίνιμουμ ε, ε, νομοθεσίες προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Ευχαριστώ κυρία Τικάου. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία και έτσι τον λόγο έχει πάλι ο Επιτροπός ο κύριος Πίμπαλης. Κύριε Πρόεδρε, κύριε και κύριοι βουλευτές, κύριε Μωρήρα αναλάβετε μια εξαιρετική πρωτοβουλία ε, για να τονίσετε το ενδιαφέρον σας για τις σχέσεις με τις, Ευρωπα... με τις Συμφωνούμε όλοι για τη σημασία των σχέσεων αυτών. Σχεδόν 2 δισεκατομμύρια ευρώ αγαθών και υπηρεσιών ε, είναι το ίσως του εμπορίου κάθε μέρα μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΗΠΑ Ενώ έχουμε και άνω των 2-3 εκατομμυρίων ευρώ σε επενδύσεις. Σχεδόν το μισό του παγκοσμίου ΑΕΠ και το 1 τρίτο του παγκοσμίου εμπορίου είναι μεταξύ των δύο ακτών του Ατλαντικού. Αυτοί οι αριθμοί δείχνουν πως η σχέση αυτή είναι μοναδική. Όμως μπορεί να γίνουν ακόμη περισσότερα. Σε καιρούς οικονομικά δύσκολους το ενισχυμένο εμπόριο βέβαια συνεισφέρει στην ανάπτυξη και στις εργασίες Γι' αυτό σκοπεύουμε η τωρινή μας πρωτοβουλία για το εμπόριο και τις επενδύσεις να επιτύχει. Στην Σύνοδο Κορυφής ε, του Νοεμβρίου 2011 συνστάθη μια ομάδα εργασίας υψηλού επίπεδου για τις δουλειές και την ανάπτυξη για να προωθηθεί το εμπόριο και οι επενδύσεις για να έχουμε αμοιβαία υποφελής επενδύσεις, οικονομική ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα. Στις 19 Ιουνίου υιοθετήσαμε μια ενδιάμεση έκθεση στην οποία καταλήξαμε σε προσωρινά συμπεράσματα για μια ολοκληρωμένη συμφωνία που θα αναφέρεται σε πάρα πολλά ζητήματα διμερούς εμπορίου η οποία βεβαίως θα ε, ήταν η καλύτερη επιλογή για τα θέματα αυτά και από πολιτική σκοπιά, καθώς επιτρέπεται έτσι να έχουμε μια λύση πακέτο. Επίσης δεν έχει ληφθεί πολιτική απόφαση. Παρ' όλα αυτά ξεκίνησε η διαδικασία στην τελευταία σύνοδο κορυφής και πηγαίνει προς αυτή την κατεύθυνση. Συνεργαζόμαστε στενά με τους Αμερικανούς συναδέλφους μας για να συντάξουμε την τελική έκθεση που μας έχει ζητηθεί πριν από το τέλος του έτους τελική έκθεση θα περιέχει συστάσεις για το τι θα γίνει από εδώ και μπρος ε, που εμείς θεωρούμε πως πρέπει να ε, είναι η έναρξη συνολικών διαπραγματεύσεων. Είναι λοιπόν επίκαιρη η έκθεσή σας ε, και συνεισφέρει στις εργασίες της ομάδας υψηλού και θα λάβουμε υπόψη τις απόψεις που εκφράσατε στο μέτρο του δυνατού. Σας ευχαριστώ και πάλι για τη συνεισφορά. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Τελείωσε η συζήτηση. Η ψηφοφορία αύριο στις 6 ώρα το απόγευμα. Επόμενο σημείο, η έκθεση της κυρίας Φώστερ για την ε, εφαρμογή της νομοθεσίας για τον ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό. Ε, τον λόγο έχει η συγγήτρια για 4 λεπτά.